Φεβρουαρίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπή υπό της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερική πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Ελευθερία έκφραση στην Τουρκία, πρόσφατα συλλήψει δημοσιογράφων, διευθυνών των στελεχών των μέσων ενημέρωση και συστηματική άσκηση πίεση ει βάρο των μέσων ενημέρωση στην Τουρκία. να ζητήσω από τον κύριο Ντελαβέντοβα να λάβει το λόγο του μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ μέρου τη ΥΠΑ, τη εκπροσώπου και αντιπροέδρου τη Επιτροπή παίρνω το λόγο και ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα η τουρκική αστυνομία συνέλαβε πολλού δημοσιογράφου και διευθύνοντα τελέχη των μέσων ενημέρωση στην Τουρκία. Όλοι παρακολουθήσαμε την είδηση αυτή με ιδιαίτερη προσοχή. Η ύπατη εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο Μογκερίνη και ο επίτροπο Χαν την Κυριακή ε, προχώρησαν σε δήλωση ε, δήλωση η οποία τονίζει χωρίς καμία αμφισημία ότι τα γεγονότα αυτά δεν συνάδουν με την ελευθεροτυπία θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας. Η δήλωση επίσης εκφράζει την ευχή ότι θα γίνει σεβαστή η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και θύμισε το παραβίαστο δικαίωμα να υπάρχει εκδίκαση διαφανής και αντικειμενική μαζί με το δικαίωμα σε συνήγορο των ε, κατηγορουμένων. Βεβαίως οι παράνομες ενέργειες πρέπει να τιμωρούνται, αλλά πάντοτε στα πλαίσια του κράτους δικαίου και με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας. Χθε το Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση και ενέκρινε σαφέστατα και αποφασισμένα συμπεράσματα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τι υποχρεώσει της Τουρκίας ως χώρας υποψηφίας στην ένταξη. Η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο ε, Επίτροπο μάλλον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Νίλ Βιουρτνέσκ, στο Συμβούλιο τη Ευρώπη εξέφρασε την ανησυχία του, ε, μιλώντα για οπισθοχώρηση σε σχέση με την ελευθερία τη έκφραση των μέσων ενημέρωση σε αυτή τη χώρα. Και το Κοινοβούλιο έκανε τη φωνή του να ακουστεί. Πολλοί ήσασταν αυτοί μαζί με τον πρόεδρο Σούλτ που εκδάσατε τι ανησυχίε σα για τι τελευταίε εξελίξει. Σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε το μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε προ την Τουρκία. Όλοι συμφωνούμε ότι η Τουρκία ως χώρα υποψήφια στην ένταξη θα πρέπει να σεβαστεί τα μέγιστα δημοκρατικά πρότυπα και ω προ τι προδιαγραφέ που ακολουθεί και τι πρακτικέ τη, με πλήρη σεβασμό τη ελευθερία έκφραση, που είναι σημαντική για να ολοκληρωθεί και να ασκηθεί μια σειρά από άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω η ελευθερία τη εισπήρωση και τη ε, διαδήλωση, όπω η ελευθερία τη σκέψη ή ε, των θρησκευτικών του πεθήσεων. δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρί αυτέ τι βασικέ ελευθερίε. Στην έκθεση του το 2014 για την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασκήψει στι θετικά βήματα πρόοδου τη χώρα αυτή, όπω το πακέτο εκδημοκρατισμού, το σχέδιο δράση κατά τη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τη Τουρκία και η πραγματική δέσμευση για να καταλήξουμε σε επίλυση του κουρδικού Ταυτόχρονα η έκθεση αυτή εξέφραζε ανησυχίες ως προς τι διάφορες εξελίξεις που φαίνεται να απειλούν ιδιαίτερα στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ελευθερία της έκφρασης τα προβλήματα ω προ την ελευθεροτυπία και την ελευθερία τη έκφραση στην Τουρκία δεν είναι καινούρια. Είδαμε τι καταστολή υπήρχε κατά των δημοσιογράφων και των κοινωνικών δικτύων μετά από τι διαμαρτυρίε στο Πάρκο Γκέτ. Επίση, με τον πρόσφατο πολιτικό διάλογο και τι διμερεί ε, συνομιλίε που είχαμε με Τούρκου εκπροσώπου, ε, παραλάβαμε ότι η διαδικασία ένταξη είναι καθοριστική σημασία για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Αλλά ταυτόχρονα εκφράσαμε και το πόσο μα απασχολεί ε, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και ε, των βασικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ιδίω τη ελευθερία τη έκφραση, διότι είναι κινητήριο δύναμη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή η πρόοδο επί τη πράξη στην Τουρκία ε, πρωτίστω για το κράτο του δικαίου και τα βασικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία ε, μαζί με τον Επίτροπο Στυλιανίδη, η ύπατη εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο Μογκερίνη και ο Επίτροπο Χάν υπογράμμισαν ότι το κράτο δικαίου και οι θεμελιώδει ελευθερίε είναι ουσιαστική τομεί όπου η AUTHORWAVE Τουρκία πρέπει να επιτελέσει πρόοδο. Όλοι οι Τούρκοι συνομιλητέ επανέλαβαν την σημασία των, σχέσεων, των καλών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχτηκαν ευνοϊκά αυτήν την κοινή επίσκεψη. Εξέφρασαν την ε, αφοσίωσή του ε, στην πορεία τη χώρα προ την Ευρωπαϊκή Ένταξη καθώ και την, ε, το πώ είναι αποφασισμένη η Τουρκία να συνεχίσει τι πολιτικέ τη μεταρρυθμίσει. Είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη και ο Επιτροπό επανέλαβαν ότι αυτή ισχυρή δέσμευση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω εκφράστηκε από του Τούρκου ομολόγου του κατά την επίσκεψή του, θα πρέπει να μεταφραστεί και σε χειροπιαστέ ενέργειε. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβαν συχνά ότι η Τουρκία είναι ένα ε, σημαντικότατο εταίρο και θεωρούν ότι πρέπει να λάβει ένα σαφέ μήνυμα ω προ την ανάγκη να γίνουν βήματα προόδου προ τι αναγκαίε προόδου με όλα τα ε, στοιχεία και τα απαραίτητα αντίτιμα για να υπάρξει εγγύηση ελευθερίας έκφρασης και ελευθεροτυπίας. Τα κράτη-μέλη επανέλαβαν ότι η διαδικασία ένταξης και προσχώρησης εξαρτώνται από το πόσο θα γίνουν σεβαστά τα θεμέλια δικαιώματα και πόσο θα ενισχυθεί το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειες της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι η διαδικασία ένταξης παραμένει το πλαίσιο αναφοράς που ενδείκνεται για να μπορέσει να προοδεύσει η Τουρκία και οι μεταρρυθμίσεις της, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό είναι πολύ σαφής και έχει ε, γίνει γνωστή και στους Τούρκους ομολόγους στόχους μας με απόλυτη σαφήνεια και συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον και οφείλει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα αυτή που είναι υποψήφια και περιμένουμε επιτέλους από την Τουρκία μια επικοδομητική δέσμευση όσον αφορά αυτές μας τις μέρημνες. Κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε καλόπιστα την πορεία της ένταξης, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαργαλεία που διαθέτουμε και η Τουρκία θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας. Εύχομαι η ευνοϊκή δέσμευση της Τουρκίας θετική δέσμευση τη Τουρκία υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει του ε, καρπού που όλοι επιθυμούμε. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, επιτρέψτε μου να σα βεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε στενά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω την συζήτηση για να ακούσω τις απόψεις σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε εκ μέρους της Αντιπρόεδρου και είπα της εκπροσώπου. Τώρα ο κύριος Πρέντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για όσα είπατε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ μιλώ σαν φίλος της Τουρκίας. Δεν είμαι από αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι έκαναν καριέρα αντιτιθέμενοι στην προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς σαν φίλος λοιπόν λέω ότι ανησυχώ και πραγματικά ανησυχώ πολύ για τις πρόσφατες εξελίξεις, τις συλλήψεις και τη γενική στάση της Τουρκίας απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται ότι η πρόθεση των Τούρκων πολιτικών είναι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Όμως είναι σαφής η πρόθεση αυτή. Και η κύρια ανησυχία, πιστεύω, είναι ότι οι επιχειρηματίες που στηρίζουν την προσχώρηση αυτή είναι αυτοί που ανησυχούν περισσότερο. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σημάδι και θα έπρεπε να προβληματίσει τις τουρκικές αρχές. Εξακολουθώ να υποστηρίζω κριτήρια για την διαπραγματεύση των κεφαλαίων 23 και 24. Είναι μια θέση που υιοθετήσαμε με το τελευταίο ψήφισμά μας όσον αφορά την πρόοδο της Τουρκίας. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω θα συνεισφέρουμε στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία γύρω από αυτό το θέμα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέλνει ένα σαφές μήνυμα αν συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με μια χώρα η οποία δεν τοποθετείται σαφώς όσον αφορά την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ίσως θα έπρεπε να συνεχίσουμε με την Μολδοβία τη διαπραγματεύσει, η οποία φαίνεται να είναι μια πιο σταθερή χώρα από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η κυρία Κάτι Πέριχη τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η διαδικασία προσχώρησης πρέπει να περάσει μέσα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αρχών. Είναι πολύ βασικό αυτό για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ανησυχούμε λοιπόν όλους ιδιαίτερως για τόσα έγιναν την προηγούμενη Κυριακή, όπου διώχτηκαν δημοσιογράφοι και συνελήφθησαν επιπλέον. Ήδη πήθηκαν επικρίσεις απέναντι στην Τουρκία, η οποία διώκει δημοσιογράφους, δεν τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα. Με τέτοια συμπεριφορά δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσει η Τουρκία. Πρέπει να υπερισχύσει η αρχή της αθωότητας εφόσον δεν έχει αποδειχθεί ενοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγα στην ε, Τουρκία ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τουρκική κυβέρνηση κατάλαβαν ότι χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Οπότε χαίρομαι από τη δήλωση που έκανε η κυβέρνηση της Τουρκίας που είπε ότι χρειάζεται επιπλέον εκδημοκρατισμός και διακανονισμός του Κουρδικού, ότι τα θέματα αυτά αποτελούν προτεραιότητα για αυτούς. Εμεί βέβαια ανησυχούμε για την επιδεινούμενη κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου στη χώρα. Αυτό όμως δείχνει ότι ακριβώς εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στη διαδικασία για προσχώρηση της Τουρκίας, αλλά τελικά είναι η τουρκική κυβέρνηση η οποία έχει τον παλάκι στο δικό της το μέρος. Εμείς εκφράζουμε ανησυχίε όσον αφορά την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν η Άγκυρα πρέπει να μας πείσει ότι εξακολουθεί να θέλει να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της. Η διαδικασία προσχώρησης είναι μοναδική ευκαιρία για την Τουρκία να αναπτύξει ένα πλουραλιστικό, ισχυρό δημοκρατικό σύστημα υπέρ όλων των πολιτών στην Τουρκία. Όμως, με τη συμπεριφορά της απέναντι στα μέσα ενημέρωσης απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό είναι πολύ κακό νέο για οποιονδήποτε είναι φίλος της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τάνοκ, ένα λεπτό. Ό,τι απόψη και να έχουμε για την πολιτική τη Τουρκική κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία ω χώρα. Από τότε που είναι υποψήφια το 2005, η διαδικασία ένταξη πάντα θα ήταν δυσχερή για μια τόσο μεγάλη και σχετικά φτωχή χώρα με πολύ διαφορετική κληρονομιά από την Δυτική Ευρώπη και νοοτροπία. Μόνο ένα κεφάλαιο το 33 έχει ανοίξει και κλείσει. για η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει τη δημοκρατία της Κύπρου. Αλλά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η επιρροή του Ισλαμιστικού ΑΚΠ και η προσέγγιση η όλο και περισσότερο πολιταρχική του Πρόεδρου Αντογάν που αντιμετωπίζει ε, που προσπαθεί να συγκρουστεί με τους πάντες το στρατό, του φοιτητέ και τώρα και άλλους Ισλαμιστές, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Και υπαναχωρεί και όσον αφορά τι διαπραγματεύσει με το ΠΚΚ και μόνο λίγο μεγάλη πίεση του ΝΑΤΟ επέτρεψε να υποστηριχθούν οι, οι κουρδικές δυνάμεις που είναι πολιορκία στο Κομπάνι. Θεωρεί ότι το κτηνόδες Ισλαμικό κράτος είναι λιγότερη απειλή παρά το ΠΚΚ και το γεγονό ότι έχουν υποστηρίξει του τζιχαντιστέ στην Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία είναι αρνητικό. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζουμε να αλλάξει πορεία η Τουρκία και να γίνει πιο φιλοδυτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σχάκε, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Όνειρο τη Τουρκία έχει γίνει ένα εφιάλτη και επιτέλου πρέπει να μπει ένα στόπ. Εγώ ήμουν από αυτού του επικριτικού φίλου τη Τουρκία που έλεγε ότι η διαδικασία τη ένταξη μπορεί να εξυπηρετεί τι μεταρρυθμίσει. Όμω πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο. Η σύλληψη των δημοσιογράφων την περασμένη εβδομάδα είναι μια διαρκή στάση τη κυβέρνηση για παραβίαση του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Τουρκία. Μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη τη ύπατη εκπροσώπου στην ε, Άγκυρα, βλέπουμε ότι οι σχέσει μα έχουν φτάσει για άλλη μια φορά στον Αδύρ. Υπάρχει υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσει και μετά τι κατηγορίε διαφθορά για τον, κύριο, κατά τον κύριο Ερτογάν που ήταν τότε πρωθυπουργό, τώρα Πρόεδρο, εκατοντάδε αστυνομικοί και ε, δικαστικοί λειτουργοί μετατοπίστηκαν και απειλήθηκαν με ε, δίκε και καταδίκε. Οι δημοσιογράφοι ήδη γνώρισαν μεγάλη πίεση στην Τουρκία. Μεγαλύτερο, το, έχει το μεγαλύτερο ρεκόρ ε, φυλακισμένων δημοσιογράφων η χώρα αυτή. Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να αντιδράσει με πυγμή. Είδαμε ότι η Τουρκία διαρκώ ολισθαίνει από τον χώρο τη δημοκρατία ε, και θα έπρεπε οι διαπραγματεύσει να πάψουν. Ωστόσο, βλέπουμε να έχουν περάσει πολλά ε, καθοριστικά χρονικά σημεία χωρί να αναλαμβάνει επιφασιστική δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την περίπτωση Αχματσέκ μέχρι τι ε, δίκε δημοσιογράφων ή με τους ε, υπερασπιστέ του Γκουλέν, που είναι ένα μόνο από τα προσπαθότερα γεγονότα σε μια σειρά από παρόμοια γεγονότα βλέπουμε να έχουν δημιουργηθεί τέρατα πλέον στην Τουρκία με ένα συνασπισμό που επιτέλους ε, ανοίγει το δρόμο για τις εξτρεμιστικές δράσεις και περαιτέρω παραβίαση του κράτους δικαίου. Σήμερα πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμού, γυναίκες, ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες Οποιοδήποτε επικρίνει την κυβέρνηση φοβούνται για τη ζωή του. Το να χάσει κανεί τη δουλειά του ή μια άδεια, το να λάβει ένα πρόστιμο από την εφορία, το να κατηγορηθεί ότι ε, έχει προσπαθήσει να ρίξει την κυβέρνηση, έχουν γίνει κατηγορίε που μπορεί να εκτοξευθούν ανα πάσα στιγμή. Και ε, όλοι απειλούνται με ε, δίωξη στη δικαιοσύνη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να δείξει ότι πρέπει να δοθεί ένα τέρμα στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αυτέ οι δράσει δεν μπορούν να συνεχιστούν επάπειρον. Ευχαριστούμε ο κύριο Χατζηγεωργίου. Το πρόβλημα που συζητάμε κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να ειδωθεί σαν ένα μεμονωμένο ζήτημα. Κάτι πάσχει στο βασίλειο της Τουρκίας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι πρόσφατες συλλήψεις. Δεν είναι μόνο η καταπάτηση τη ελευθερία του λόγου είναι τα διατρέξαντα στο πάρκο γκεζί είναι η στάση της τουρκίας στο κομπάνι είναι η στάση της τουρκίας απέναντι στο κουρδικό είναι η στάση της χώρας απέναντι στην κύπρο το κάζους μπέλι κατά της ελλάδας είναι η στάση απέναντι στις γυναίκες και στις μειονότητες είναι η στάση του κυρίου ερντογάν στάση απαξίωσης απέναντι στις αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου μια στάση που λέει πως τα ψηφίσματά μας θα πάρουν την άγουσα για τον κάλαθο των αχρήστων εμείς ως Κύπριοι ευρωβουλευτές καθόλου δεν χαιρόμαστε γι' αυτά. εμείς θέλουμε μια γείτονα χώρα δημοκρατική μια χώρα που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα τους γείτονές της και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. πιστεύω απόλυτα πως πρέπει η τουρκία να πάρει καθαρό και σκληρό μήνυμα από την ευρωπαϊκή ένωση και καθαρό μήνυμα σημαίνει κυρώσεις για τη συμπεριφορά της. οι και τα χαϊδέματα δεν θα βοηθήσουν καθόλου. είτε θα κατανοήσουν ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν είτε θα συνεχίσουν το δούλεμα. είμαι βέβαιος ότι χωρίς αυτό το μέτρο το μέτρο των κυρώσεων και αυτή η συζήτηση και το πιθανό ψήφισμα που θα ακολουθήσει θα πάρει τον γνωστό δρόμο του καλάθου. καθαρό μήνυμα σημαίνει κυρώσεις αλλά σημαίνει και ειλικρίνεια εκ μέρους μας για την ενταξιακή της πορεία. σας καλώ να χαλιναγωγήσουμε αυτή την άδικη συμπεριφορά. σας καλώ να υψώσουμε ανάστημα απέναντι στο χαλιφάτο του κυρίου Ερτογάν. Και τώρα δύο λεπτά η κυρία Χάρμς. Να πω κάτι ευθύ εξ αρχής. Πρέπει όλοι σε αυτή τη συζήτηση να καταστήσουμε σαφές κάτι ότι κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση Νταβουτόγλου και στον πρόεδρο Ερντοάν ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσεις στα σύνορα της Τουρκίας, τον πόλεμο στη Συρία και το Ισλαμικό κράτος. Αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε από κοινού καθώς και την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή των προσφύγων, τη χιονοστιβάδα των προσφύγων σε αυτή την περιοχή. Αυτό να μην το ξεχάσουμε στη συζήτηση που κάνουμε, γιατί είναι κοινή πρόκληση αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι σωστό ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι αυτών που συνέβησαν τον προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Οι συλλήψεις και οι διώξεις κατά δημοσιογράφων, αστυνομικών και οι έρευνες σε εφημερίδες και σε σπίτια που ε, έχουν ήδη συμβεί και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν εάν εμείς δεν τα καταγγείλουμε έντονα. Η κυβέρνηση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρεί ότι όλες οι δραστηριότητες της αντιπολίτευσης, όλες οι επικρίσεις, και αυτό δεν είναι μόνο το κίνημα Γκουλέν και τα μέσα, όλες οι δραστηριότητες ε, που την επικρίνουν θεωρεί ότι είναι συνωμοσία ανατροπής του κράτους ή συνωμοσία προετοιμασία πραξικοπήματο κατά του Πρόεδρου Αντοάν και της πλειοψηφία του. Αυτό θεωρώ είναι απόλυτα αδιανόητο. Οι διαμαρτυρίε, για παράδειγμα και οι διαδηλώσει στο Γκεζί, οι διαδηλώσει κατά του Ισλαμικού κράτους, οι διαδηλώσει ε, για τα θύματα του Κομπάνη και τα μνημόσυνα. Όλα αυτά θεωρούνται ως τμήμα μιας τεράστιας συνωμοσία. Εάν θέλουμε να επικρίνουμε αυτό που συνέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τότε πρέπει συνολικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που συχνά τίθεται μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης και επίσης και μεταξύ κυβέρνησης και μειονοτήτων. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε επίκριση θεωρείται έκκληση για πραξικόπημα και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Βίνμπεργκ έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Τουρκία για άλλη μια φορά παραβιάζει την ελευθερία έκφρασης και οι επιθέσεις της στα μέσα ενημέρωσης την εκθέτουν. Καμία χώρα δεν κατέφυγε στα δικαστήρια τόσο συχνά για να πνίξει την ελευθερία έκφρασης ως η Τουρκία. Παρά τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αλλάξει στάση η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια διαμαρτύρεται κατά της ε, συνεχιζόμενης αυτής ε, βίας στην οποία εκτίθενται οι πολίτες, οι Τούρκοι. φυλακίσεις επαναλαμβανόμενες. σε 66 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε με δημοσιογράφος πρόσφατα και άλλοι επίσης. Σε 6 χρόνια φυλάκιση. Δημοσιογράφοι από το Λατάς, για παράδειγμα, από το Γαλατά πολλές φορές καταδικάστηκαν. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πάνω από 900 εκατομμύρια πήγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Τα χρήματα αυτά τα πήρε η Τουρκία ως αντάλλαγμα για την βελτίωση που διαπιστώθηκε σε θέματα ασφάλειας για να αποφεύγεται η διαφθορά και για να τηρείται το κράτος δικαίου. Δεν επενδύσαμε όμως καλά από ό,τι φαίνεται. Για μένα μου η Τουρκία δεν θα ανταποκριθεί ποτέ στις προδιαγραφές μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Σαλβίνη 1,5 λεπτό. Έκομαι. Να με. Είναι απίστευτο ότι από 15 χρόνια επιμένουμε να θέλουμε να εντάξουμε την Τουρκία στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα κράτος που κατέχει εδώ και 40 χρόνια το τμήμα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, με στατιωτικά μέσα. Έχουν καταστρέψει εκκλησίες και έχουν ε, κάνουν κατοχή των εδάφων. Έχουν προχωρήσει η γενοκτονία των ε, Αρμενίων, ένα εκατομμύριο ε, νεκροί. Και θυμηθείτε τι σφαγή υπήρξε με την αφορμή της επαιτίου αυτά τα Χριστούγεννα. Επίσης δεν μιλάμε απλώς για ένα κράτος που παραβιάζει τα δικαιώματα των δικαιωμογράφων, των δημοσιογράφων. Μιλάμε για ένα κράτος που δεν θα γίνει ποτέ Ευρώπη, στις εμπορικές, στις στατικικές, στις οικονομικές μας σχέσεις. Συνεχίζουμε να τους δίνουμε όμως λεφτά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τους πληρώνουμε ένα κράτος που κατέχει εδώ και 40 χρόνια ένα άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνωρίζει ότι σφαγίασε ένα εκατομμύριο ανθρώπου και τον επόμενο Απρίλιο γιορτάζεται η εκατονταετρίδα από την γενοκτονία των Αρμενίων. Εδώ, σε αυτό το μέγαρο θα θυμηθούμε το, την εκατονταετρίδα από την γενοκτονία των Αρμενίων και τους δίνουμε 100 εκατομμύρια το χρόνο. Ε, η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνουμε στο χέρι 100 εκατομμύρια, cash, 100 ε, εκατομμύρια και του χρόνου, 100 εκατομμύρια και σε δύο χρόνια και σε τρία. Και εκείνοι τι κάνουν, ε, ξοδεύουν τα λεφτά μας για να κάνουν θέματα ανταγωνισμού στι επιχειρήσει μα και να συλλαμβάνουν δημοσιογράφου. Η Τουρκία δεν θα είναι ποτέ Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον το πούμε για να είμαστε σοβαροί. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Σαλβίνη, ε, έχει ζητηθεί μια ερώτηση με μπλε κάρτα από τον κύριο Μπενιφέη. Το αποδέχεστε? Ωραία, έχει 30 δευτερόλεπτα ο κύριο Μπενιφέ για να σας ε, θέσει την ερώτησή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να μου πει ο κύριο Σαλβίνη, εάν θεωρεί ότι αυτά που είπε για την Τουρκία μπορεί να ισχύουν και για την Ρωσία του, του, του Πούτιν. Μιλήσατε για κατοχή εδαφών. Για θυμηθείτε την κατοχή της Κρυμαίας, την παράνομη εισβολή εκεί, τη συμμετοχή στις συγκρούσεις στα ανατολικά της Ουκρανίας. Μιλήσατε για παραβίαση δικαιωμάτων. Τι γνώμη έχετε για τη Ρωσία επ' αυτών. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαλβίνη. Φαντάζομαι ότι κάνατε πλάκα Νομίζω ότι το λέτε για αστείο, έτσι. Στην Κρυμαία ψήφισαν. Υπήρξε δημοψήφισμα και το 95% των πολιτών ε, με την παρουσία διεθνών παρατηρητών αποφάσισαν ότι αυτή την πορεία θα πάρει η Κρυμαία. Ε, νομίζω ότι η παρέμβαση του συναδέλφου ήταν μια συμπαθητική πρόκληση πρώτων Χριστουγέννων και μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία δίνουμε 100 εκατομμύρια το χρόνο. Στη Ρωσία χαρίζουμε οικονομικέ κυρώσει που του έχουν γονατίσει. Και αυτό είναι και αντίθετο με τα συμφέροντά μα. Το παίρνω λοιπόν για πλάκα και αποφεύγω να απαντήσω. Ε, Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ζόμερ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι περιορισμοί της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία δεν είναι καινούριο χρόνια τώρα. Όσοι επικρίνουν ε, αναγκάζονται να σιωπήσουν, φυλακίζονται με αντιτρομοκρατικούς νόμους. Είναι γελιογραφία η κατάσταση. Τα κοινωνικά μέσα επίσης ε, τα κλείνουν. Και τώρα έχουμε και νέες επιδρομές και τις συλλήψεις της ε, προηγούμενης Κυριακής. Αυτό φυσικά ε, δεν είναι σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αξίες μας. Η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης είναι αδιανόητο να παραβιάζονται σε μια δημοκρατία. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Και αντί για αυτές τις ελευθερίες βλέπουμε τόσο αυθαίρετους περιορισμούς και μια τέτοια χώρα ποτέ δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ένωση. Ωστόσο, η Τουρκία η Τουρκία και κανένα άλλο βασικό πολιτικό κριτήριο δεν ε, τήρει για παράδειγμα οι προσπάθειες αντιμετώπισης της διαφθοράς ε, μελών της κυβέρνησης και άλλων μελών της ε, πολιτικής ελίτ. Βλέπουμε ότι παρεμβαίνουν στις ε, έρευνες και οι δικαστές και οι αστυνομικοί που προσπαθούν να ερευνήσουν τέτοια φαινόμενα απολύονται, μετατίθενται. Διότι έτσι θέλει ο πρόεδρος Ερντοάν, γιατί ε, έχει κατηγορηθεί και ο γιος του. Άρα κράτος δικαίου δεν υπάρχει στην Τουρκία. Μόνο η αυθαιρεσία του πρόεδρου Ερντοάν. Η χώρα λοιπόν αυτή οπισθοδρομεί τρομερά και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αφελείς επιτέλους έναντι της χώρας αυτής. Να σκεφτούμε τι κυρώσεις μπορούμε να επιβάλλουμε. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου κάνω έκκληση στο τουρκικό συνταγματικό δικαστήριο να προσπαθήσει να σταματήσει αυτές τις εξελίξεις. Τέτοιες χονδροειδείς παραβιάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρίτσαρτ Χάουιτ. Τώρα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κανείς δεν είναι ασφαλής στην Τουρκία σήμερα. Αυτά λένε οι αρμόδια τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους οποίους μίλησα στο τηλέφωνο νωρίτερα σήμερα. Δυστυχώς ο αριθμός των δημοσιογράφων και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που διώκονται και βρίσκονται στη φυλακή είναι κάτι ασύμβατο με τη δημοκρατία. Οποιοςδήποτε είναι κατά της κυβέρνησης φυλακίζεται. Είναι πράγματα ιδιαίτερα ανησυχητικά και τίθενται πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη δικαστική εξουσία. Υπάρχουν κατηγορίες για τρομοκρατικές οργανώσεις. Πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η Τουρκία έχει προβλήματα με τον νόμο κατά της τρομοκρατίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, από ό,τι μου λένε οι ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν τηρούνται, φυλακίζονται, διώκονται άνθρωποι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτά βέβαια τετίθενται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. θα έπρεπε να υπάρξουν ε, διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία έχει πάρει το δρόμο του κράτους δικαίου. Αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Η νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας δεν είναι όπως θα έπρεπε. Οι δημοσιογράφοι καταλήγουν να συλλαμβάνονται και πρέπει εκείνοι να αποδείξουν την αθωότητά τους. Η Τουρκία μπορεί να μιλάει για το κράτος δικαίου, αλλά στην πραγματικότητα δεν το τηρεί. Τέλος, Πρόεδρε. Όσοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά για να μιλήσουν κατά της προσχώρησης της Τουσκίας, για μένα το μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι πρέπει να δεσμευτούμε ακόμα περισσότερο υπέρ της Τουρκίας, να τη βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Βέβαια η συγγήτρια πρέπει να κάνει τη δικιά της τη δουλειά για την έκθεσή της όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία όμως είναι μια χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουμε όπως και τους Τούρκους. Υπάρχουν δύο μπλε κάρτες για σας. Ο κύριος Τάνοκ πρώτα και ο κύριος Φαντούλης ο δεύτερος. Δέχεστε. Ο κύριος Τάνοκ πρώτα. Έχετε τη φήμη ότι είσαστε φίλος της Τουρκίας, πράγματι, και στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα να σας ακούω σήμερα, να είσαστε επικριτικός δηλαδή όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αν συνεχιστούν αυτές οι παραβιάσεις εδώ θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα χρήματα των φορολογούμενων που πηγαίνουν στην Τουρκία και τη χρηματοδοτούν. Αλλιώς τι κυρώσεις μπορούμε να επιβάλλουμε σε μια υποψήφια για προσχώρηση χώρα. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον δεύτερο ερωτώντα, και μετά στον κύριο Χάγη να απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. Ο κύριος Φουντούλης, παρακαλώ. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας, αφού εκφράσατε τη γνώμη σας για την Τουρκία που όλοι ξέρουμε ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διώκονται η πολιτική σκέψη, ποια είναι η γνώμη σας για τις διώξεις που γίνονται στην Ελλάδα εναντίον του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή και ο αρχηγός μας και οχτώ βουλευτές βρίσκονται προφυλακισμένοι με ανυπόστατες κατηγορίες και είναι τόσο υποκριτικό ότι κανείς από εδώ μέσα δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Χάουιτ ένα λεπτό για να απαντήσει. Κύριε Φουντούλη, συμφωνώ απόλυτα ότι όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταδικάζονται ισότιμα. Αλλά αυτό που με ανισχύει για τη συζήτηση εδώ είναι ότι άκουσα πάρα πολλούς που σπρώχνονται για να καταδικάζουν την Τουρκία, αλλά για άλλες χώρες όπου η κατάσταση είναι ίδια ή χειρότερη δεν το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς. Πρέπει να υπερασπιζόμεθα παντού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο φίλο μου τον κύριο Τάνοκ, πρώτα απ' όλα του λέω καλά Χριστούγεννα. Βεβαίω, σωστά μπορούμε να πούμε ότι ναι, μεν είμαι φίλο τη Τουρκία και με χαρά δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Αγαπώ τη χώρα αυτή και θέλω να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω να γίνονται εκεί. Είναι σωστό να πούμε ότι έχει διαφορετική αντίληψη από μένα. Και θα συνεχίσει να έχει αυτή την άποψη και θα την είχε και πριν το Σαββατοκύριακο. Και το συζήτησα σήμερα με τον αρμόδιο επίτροπο και είπα ότι δεν θέλουμε προληπτικέ ενέργειε σε σχέση με την ένταξη. Και ο επίτροπο Χάν μου είπε ότι συμφωνεί μαζί μου να καταδικάσουμε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, αλλά α σκεφτούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσερμιτ. Μέσερμιτ. Μα κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι διάκριση να, ευχα... Ε, να εύχεστε καλά Χριστούγεννα μόνο στον κύριο Τάνο. Πρέπει να ευχηθείτε σε όλους. Και τώρα να δώσω στον κύριο Μέσονη το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κάποιε φορέ μερικέ κυβερνήσει φαίνεται ότι μπορούν να κοροϊδεύουν κάποιου πολίτε μερικέ φορέ και ίσω όλου του πολίτε, μερικού πολίτε όλε τι φορέ. Αλλά δεν μπορεί να ε, ισχύει αυτό συνέχεια όπω κάνει η κυβέρνηση τη Άγκυρα. Δεν μπορεί να εξαπατώνται οι πολίτε τη Τουρκία πιστεύοντα ότι μπορούν να γίνουν πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν σέβεται η χώρα αυτή κανένα από τα δικά μα κριτήρια. Δεν μπορεί να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντα να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης με όσα τώρα γίνονται. Βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει πάρει τελείως την αντίθετη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την πορεία της προς την Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε κάθε λόγο να αναζητούμε εναλλακτικέ και να δώσουμε ένα τέρμα στη δικασία των διαπραγματεύσεων. Α το σκεφτούμε επιτέλου. Μια τεχνική συνεργασία, μια συμφωνία ελεύθερου εμπολίου για τι ανταλλαγέ. Κάτι. Αλλά είναι τελείω μη ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένταξη στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε ο κ. Λιαρίκ για Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, για τα όσα έγιναν στην Τουρκία την περασμένη ε, Κυριακή πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο μία διάκριτη επίθεση κατά των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και κατά του Εβραίου κοινού. Με, 13, ε, με σε 13 τουρκικέ πόλει ε, δημοσιογράφων και διευθυντών τηλεοπτικών καναλιών. Εδώ μιλάμε για ανθρώπου που ε, αντιλέγουν στο και κατακρίνουν την πολιτική διαφθορά τη κυβέρνηση 150 οι δημοσιογράφοι απειλήθηκαν με σύλληψη μέχρι το τέλος του μήνα. Και οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να είναι αποφασισμένες και κάθετες κατά των ε, ε, σοβαρότατων αυτών παραβιάσεων των θεμελιωδών ελευθεριών. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς αυτές και κύριε Υπουργέ, εξονόματος του Συμβουλίου, δεν μπορείτε να δεχτείτε το θάνατο, την, δεν μπορείτε να δεχτείτε το νεκροτομείο που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ορντογάν. Πρέπει να αφήσουμε τους ε, δημοσιογράφους ελεύθερους για να ασκήσουν ε, την ε, ελευθεροτυπία που είναι το αντικείμενό τους με την παρέμβαση των τουρκικών αρχών στον δικαστικό τομέα ε, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά εάν ε, οι εμπορικέ μα προτεραιότητες στην εξωτερική μα πολιτική θα περνάνε μπροστά από, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα του να ενημερώνεται κανεί και να ενημερώνει, την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. και αν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοιε δράσει, ώστε κράτη που θεωρούμε εταίρου μα, να μην σέβονται τα βασικά δικαιώματα διότι δεν μπορεί το δικαίωμα της ανθρώπινης ζωής να περνά πάνω από τα να μένει μετά τα δικαιώματα των αγορών. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Τουρκία δεν είναι παρά μία όχι πολύ καλά καλυμμένη επίθεση κατά του τύπου για τις ελευθερίες έκφρασης. Οι δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται με παράλογες κατηγορίες και τους απευθύνονται κατηγορίες και φυλακίζονται και αυτοί που είχαν συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις Γκεζή κατηγορούνται τώρα για απόπειρα πραξικοπήματος. Και η αστυνομία που είχε ασκήσει βία εναντίον τους δεν έχει πάθει τίποτα. Ο Ερντοάν, από ό,τι φαίνεται, θεωρεί ότι κάθε επίκριση εναντίον του πρέπει να καταπνιγεί. Αλλά αυτό είναι το αντίθετο από κάποιον που θέλει να υπάρχει δημοκρατία. Η Τουρκία μπορεί από μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών και από ένα ζωντανό και κριτικό τύπο μόνο να υποφεληθεί. Χωρίς κράτος δικαίου και δημοκρατικές προδιαγραφές η Τουρκία ποτέ δεν θα προχωρήσει. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώς τα κράτη-μέλη έχουν κάνει και αυτά λάθη. Διότι κάποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν πάντα τη διαδικασία ένταξης και ε, κλείνουν κεφάλια λέγοντας ότι και να κάνει η Τουρκία ποτέ δεν θα τη δεχτούμε. Αυτό δεν βοηθάει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, δεν βοηθάει τις επικριτικές φωνές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τώρα μοχλό για να πιέσουμε την Τουρκία. Ε, στην ουσία βάζουμε τα χέρια μας και βάζουμε τα μάτια μας. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Σε μια διαδικασία ένταξης πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη να είναι ε, στην πρώτη γραμμή πολύ περισσότερο από τα θέματα των οικονομικών σχέσεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κάρβερ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ενώσω τη φωνή μου όσου καταδικάζουν την άδικη συμπεριφορά τη Τουρκία και τους, τις δημοσιογράφων. Με τόσε προσπάθειες να θυμωθεί η ελευθεροτυπία ο πρόεδρο Ερντογάν και το κόμμα του, ε, των οποίων ένα από τα μέλη καταδίκασε την ελευθερία των γυναικών να μπορούν να γελάνε στον δρόμο, να κυκλοφορούν ελεύθερα, ε, είναι βεβαίω κάτι που είναι απαράδεκτο για του Βρετανού συντηρητικού. Ε, το ελληνικό κράτο Τουρκίας, αυτό που δημιούργησε ο Κεμάλα τα Τούρκ, ε, είναι κάτι που έχει παραβιαστεί πλήρως. Θα πρέπει να τρίζουν τα κόκαλα στον τάφο του. Ε, στο, στη χώρα μου μόνο το UKIP ε, διαφωνεί με την ένταξη της Τουρκίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 83 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες θα έπρεπε να κυκλοφορούν ελεύθερα, αλλά αυτό έχει γύρει συζητήσεις περί μετανάστευτης στη χώρα μου. Έχει οδηγήσει σε μια ε, αντιπαράθεσή μας με τους δημοκρατικούς, του εργατικού και τους φιλελεύθερους στη χώρα. Θα έπρεπε οι πολίτες τη Τουρκία να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα προς τις χώρες μας για να αναζητούν εργασία με 9,8 εκατομμύρια ανέργους, με οποιαδήποτε μεταναστευτική ροή να επιβαρύνει τα προβλήματά μας σε τέτοιες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τουρκία λοιπόν με 1,6 πρόσφυγες πολλούς από τη Συρία και το Ιράκ τι θα γινόταν ως νέο κάτω μέλος. Μία δίωδος για την Ευρώπη για ένα ε, αριθμό προσφύγων και μεταναστών από τη Μέση Ανατολή. Πώς θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε αυτούς τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθερα με ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Οι αποσχέσεις λοιπόν ε, των, των Ευρωπαίων Υπουργών για ένταξη Τουρκίας είναι ε, αυταπάτες. Ε, ας ευχηθούμε λοιπόν τουλάχιστον καλά Χριστούγεννα και καλή Χάνουκα. Πρώτο σκεφτούμε τέτοια θέματα. Συνάντηνος. Τώρα κύριο Συνάδινος, ένα λεπτό. Πρόσφατα ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από την Ευρώπη. Κάποτε ένας γεωργός το χειμώνα βρήκε ένα παγωμένο φίδι, το σπλαχνίστηκε, το πήρε και το έβαλε στον κόρφο του. Το φίδι κάποια στιγμή αφού ζεστάθηκε και συνήλθε τσίμπησε τον ευεργέτη του. ξεψυχώντας εκείνος είπε «καλά να πάθω αφού λυπήθηκα ένα κακούργο». το προαναφερθέν παραμύθι είναι από τους μύθους του εσώπου. ανταποκρίνεται όμως πλήρως στη σημερινή πραγματικότητα. φανταστείτε την ευρωπαϊκή ένωση ως γεωργό και την τουρκία ως φίδι και σκεφτείτε πόσο ανόητο είναι η προσπάθεια προσέγγισης με την τουρκία και η ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. μια χώρα άκρως απολυταρχική που δεν σέβεται τα δικαιώματα ανθρώπων και κρατών και αγνοεί αποφάσεις διεθνών οργανισμών. μην εκπλήσεστε λοιπόν με την έλλειψη ελευθερίας έκφρασης στην τουρκία και τις διώξεις μέσων και δημοσιογράφων. ακόμα δεν έχει στεγνώσει το αίμα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην πλατεία ταξίμ της κωνσταντινούπολης. ρωτήστε διαβάστε ερευνήστε και συνειδητοποιήστε. παράνομη εισβολή και κατοχή μέρους της κύπρου χώρας μέλους ευρωπαϊκής ένωσης και επίδειξη επιθετικότητας στην αός αυτής γενοκτονία των ποντίων και αρμενίων πογκρόμ διώξεων των κούρδων προσπάθεια εκτουρκισμού και εξισλαμισμού στο τόξο βοσνία αλβανία φύρομ βουλγαρία ανοχή και παροχή βοήθειας προς τους εγκληματίες του ισλαμικού κράτους. πρέπει να κατανοήσετε ότι με την ανοχή που επιδεικνύεται προς τις τουρκικές συμπεριφορές ενισχύεται και εκτρέφεται την τουρκική προκλητικότητα και τον αυταρχισμό της. Ε, ο κύριος Χόκμαρκ έχει τώρα το λόγο. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα και είναι απλό. Η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να ελευθερώσει όλους τους δημοσιογράφους και να σταματήσει να τα βάζει με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να γίνει, ό,τι και να πούμε για το μέλλον της Τουρκίας στην Ευρώπη είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρόκειται και για τις προϋποθέσεις που ζητάμε από όλες τις χώρες να σέβονται το κράτος δικαίου και την ελευθερία έκφρασης. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να στηρίξουμε τη, μια τέτοια εξέλιξη. Να μπορέσει η Τουρκία δηλαδή να γίνει μια σύγχρονη κοινωνία με κράτος δικαίου. Μια ανοιχτή, δημοκρατική κοινωνία με ίδια δικαιώματα για τους άντρες και τις γυναίκες. Αυτή είναι η Τουρκία για την οποία θέλουμε να μιλάμε στο μέλλον προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν συζητήσαμε για τη σημερινή Τουρκία. Δεν είπαμε ποτέ ότι η σημερινή Τουρκία θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι λόγοι είναι διάφοροι. Ορισμένε χώρε προσπάθησαν να κλείσουν την πόρτα. Ορισμένοι Τούρκοι πολιτικοί επίσης μπορεί να θέλουν να κλείσουν την πόρτα. Ο κύριος Ερτογκάν στρέφει την χώρα του προς τη λάθος κατεύθυνση. Όχι μόνο την απομακρύνει από την ένταξη, αλλά την απομακρύνει και από μια σταθερή και ανοιχτή κοινωνία. Εμείς πρέπει να ζητήσουμε αλλαγές στην Τουρκία. Και κύριε Πρόεδρε, τήρησα το χρόνο μου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Βαλινθιάνο έχει τώρα το λόγο. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Χόκμαρ, προηγουμένως υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Συμφωνείτε? Ο κύριος Μαλτέζε θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ κύριε Μαλτέζε. Εγώ προέρχομαι από την Κύπρο. Είμαι Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής και είμαι από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου σας ρωτώ ευθέως με όσα έχει κάνει η τουρκία μέχρι σήμερα και δεν αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία αν ήταν η δική σας η χώρα η κυπριακή δημοκρατία θα ανεχόσασταν να μην σας αναγνωρίζει μέχρι σήμερα θα ανεχόσασταν όλα αυτά που κάνει και για να μην παρεξηγηθώ είμαι ο πρώτος που θέλω να έχει ευρωπαϊκή προοπτική η τουρκία για να επιβιώσουμε εμείς. αν για σας αυτό είναι πολιτικό όραμα για μας είναι θέμα επιβίωσης. Απαντήστε στο ερώτημα όμως για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, ναι, να απαντήσω. Βεβαίω, Το θέμα του διχασμού της Κύπρου πρέπει να λυθεί. Και αυτό αποτελεί μέρος των όσων πρέπει να γίνουν με διαμεσολάβηση και πολιτικές συμφωνίες, ώστε να είναι εφικτό στη συνέχεια η Τουρκία να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας δούμε και τα γεγονότα ότι η Τουρκία που προσανατολίζεται προς την Ευρώπη και κάνει τα σωστά πράγματα θα κάνει το σωστό και για την Κύπρο. Ενώ μια Τουρκία η οποία στρέφεται αλλού προς τη Ρωσία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού δεν θα κάνει τα σωστά. Οπότε έχουμε κοινό συμφέρον να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να στηρίξουμε σωστές και καλές εξελίξεις στην Τουρκία γιατί είναι προς όφελος της ίδιας της Ευρώπης.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 Αρχίζω και πάλι. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έλεγα ότι οι δράσεις που έχουν γίνει κατά των δημοσιογράφων και του τύπου στην Τουρκία πρέπει οπωσδήποτε να καταδικαστούν. Όπω ε, συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, που το καταδικάζουμε όχι μόνο για την ε, επιθέση κατά τη ελευθερία έκφραση, αλλά γιατί αποστελούν ένα μήνυμα που ε, δείχνει ότι δεν μα αρέσει ο τρόπο με τον οποίο οδηγεί ο Ερδογάν τη χώρα του και η κατεύθυνση στην οποία την κατευθύνει και κυρίως ο λόγος της κυβέρνησης γίνεται όλο και πιο μυσαλόδοξος. Η σοσιαλιστική ομάδα στο, στην αίθουσα αυτή και κυρίως οι Ισπανοί σοσιαλιστές πάντα υποστηρίξαμε την ανάγκη η, Ευρωπαία, η Τουρκία να έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ε, χώρο συνεννόηση για κάτι που θα ήταν καλό και για την Τουρκία και για την Ευρώπη, για όλε τι περιοχέ του κόσμου που είναι σημαντικέ για την ε, σταθερότητά μα. Αλλά γι' αυτό η τουρκική κυβέρνηση πρέπει από την πλευρά τη να κάνει αυτό που τους αναλογεί και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την βούλησή της ε, να προχωρήσει σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί τώρα τελευταία μας έχουν δημιουργηθεί πολλές ε, αμφιβολίες. Κάθε αδίκημα πρέπει να διώκεται, αλλά στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Και παρακολουθούμε πολύ κοντά τις ενέργειες του Ερντογάν. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Τουρκία, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα, λόγο, για λεπτό λοιπόν έχει το λόγο ο κύριος Δεμεσμάκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον Ιούνιο πέρυσι συνάδελφοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησαν ψήφισμα για τη σκληρή στάση της Τουρκίας απέναντι στους πολίτες στο πάρκο Γκεζή. Και εμείς καταδικάσαμε βέβαια την έλλειψη ελευθερίας ε, τύπου στην Τουρκία. Βελτιώθηκαν τα πράγματα, όχι. Αντίθετα, υπάρχει βία σε βάρος δημοσιογράφων από πλευράς του κράτους της Τουρκίας που οδηγεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί οι κανονικά δημοκρατικές χώρες σέβονται πάντα την ελευθερία έκφρασης, κάτι το οποίο δεν γίνεται εδώ. Αντίθετα, για μένα αυτή η ελευθερία είναι εγγύηση για αντικειμενικότητα όταν μιλάμε για δημοσιογράφους. Δυστυχώς όμως οι Τούρκοι συνάδελφοι υποφέρουν και με το άλοθη της εθνικής ασφάλειας συλλαμβάνονται και καταδικάζονται. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό σημάδι. Η Άγκυρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετικό δρόμο και δεν σέβεται αυτό που εγώ θα ονόμαζα νοσοποιητικό σύστημα που είναι ελευθερία έκφραση σε μια δημοκρατία. Δυστυχώς όμως πρόκειται για ένα προσωπείο που έχει η Τουρκία όσον αφορά τη δημοκρατία και πίσω από αυτό η Τουρκία αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Διακόπτεται ο μιλητής από την Πρόεδρο. Ο κύριος Μαρτέζε. Πρόεδρε, νομίζω από τη συζήτηση αυτή προκύπτει ότι με τις παρεκτροπές της κυβέρνησης Ερντογάν φαίνεται ότι και εμείς πρέπει να βάλουμε κατά μέρος την υποκρισία και τις αμφιβολίες μας. Έχουμε μια χώρα ε, με το ρεκόρ φυλακισμένων δημοσιογράφων, εκατοστή πεντακοστή ε, από την ε, κατάταξη της Σαν ε, και καταλήγει ακόμα και πιο χαμηλά όσο περνάει ο καιρός. Μιλάμε για δημοσιογράφους που ε, το κίνημα του κυρίου Γκουλέν. Οποιαδήποτε θρησκευτική κίνηση αριστεράς, δεξιάς, υπέρ των Κούρδων κατα... φαίνεται να καταστέλλεται, διότι στην Τουρκία πλέον πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα και ένα απλό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ένα επάγγελμα που εγώ ασκώ εδώ και 35 χρόνια για την διαφθορά, θεωρείται από την κυβέρνηση και τις αρχές ή την αστυνομία ω τρομοκρατική ενέργεια. Ακόμη όμω και το είδο αντίδραση, τη υπεροπτική αντίδραση του Προέδρου Ερδογάν στις ε, επικριτικά σχόλια των επιτρόπων μας ε, και τη ΥΠΑ εκπροσώπου, του κ. Χάνη και τη κ. Μογκερίνη, δείχνουν ότι η πολιτική τη Ένωση προ την Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι μια πολιτική εσφαλμένη, διότι του βοηθήσαμε να γίνουν πιο δημοκρατικοί με αυτό το σύστημα επιδοτήσεων, βοηθειών, ε, διαπραγματεύσεων. Όχι. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να φανούμε αποφασισμένοι απέναντί του. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ω τώρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, τελείωσε ο χρόνο σα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαραγκάλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ακριβώ από ένα χρόνο προέκυψε μια σοβαρή περίπτωση διαφθορά στην Τουρκία διαφθορά σε πολύ ψηλό επίπεδο πριν από μερικές μέρες, ώρες μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο του νόμου για την ασφάλεια, υπήρξε μια εκτεταμένη αστυνομική δράση κατά ενό συγκεκριμένου ε, ομίλου ΜΜΕ και κατά πρώην αστυνομικών τη αστυνομία όλα αυτά είναι απαράδεκτα σε σχέση με τη στάση που θέλει να δείξει η Τουρκία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφή άποψη, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ τη ε, κοινωνία και αυτά τα οποία κάνουν ορισμένε τουρκικέ αρχέ που είναι αντίθετε με οποιαδήποτε προσπάθεια να προχωρήσουν οι προγραμματεύσει ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν για λόγους φιλίας με την Τουρκία. Να προτείνουμε πρώτον να ζητήσουμε από τον Τούρκο Υπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις να έρθει αμέσως ενώπιον της Μικτής Επιτροπής για να μας ενημερώσει για το τι συνέβη. Δεύτερον, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την ένταξη και να ανοίξουμε γιατί όχι τα κρίσιμα κεφάλαια 23 και 24 ακριβώς για να εκφράσουμε στα πλαίσια αυτά περισσότερες ανησυχίες για αυτές τις ε, ενέργειες. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Κοράου, 1,5 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μια επίθεση ανάλογη των ε, απολυταρχικών κρατών ε, συνέλαβε 24 δημοσιογράφους ε, η τουρκική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα επειδή επέκριναν την κυβέρνηση Ερντογάν για τις περιπτώσεις διαφθοράς στην Τουρκία. Πρόκειται για κάτι που παραβιάζει όλες τις αρχές ελευθερίας έκφρασης οι οποίες θεμελιώνουν κάθε δημοκρατία. Ήδη καταπολεμάται κάθε προσπάθεια αντιπαράθεσης στο επίσημο καθεστώς. Μιλάμε για μια σειρά από καθημερινές παραβιάσεις για οικονομικές για οικονομικέ ατασταλίε που επικρίνονται για τα μέλη τη οικογένεια του ίδιου του Προέδρου τη Τουρκία, ε, με μια αστυνομία που δεν ασκεί τα καθήκοντά τη και το δικαστικό λειτουργήμα να είναι στα χέρια των πολιτικών. Και βεβαίω με το μεγαλύτερο αντίπαλο του Ερντογάν, τον Γκουλέν, να, να καταδιώκεται. Επίσης το Twitter και το YouTube ε, διώκονται διότι θεωρούνται μέσα ε, ε, για τη διάδοση των τάσεων των αντιφρονούντων όπως εκφράστηκαν στην πλατεία Ταξίμ και στο Πάρκο Ε, Ο Ερντογάν λοιπόν με τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτηκε να βρει και να απαντήσει μόνο μία, με μια επιρροπτική δήλωση. Κοιτάξτε τη δουλειά σας. Αυτό παραβιάζει όλες τις ευρωπαϊκές αξίες και τα πρότυπα της Ένωσης που η Τουρκία ίδια φιλοδοξεί να ε, στην οποία φιλοδοξεί να συμμετάσχει. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί τέρμα στις ανταδικαιματικές τάσεις είναι οι οικονομικές κυρώσεις. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριο Φεράν. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζονται περισσότερα. Βλέπετε, τι άλλο χρειάζεστε μάλλον για να δείτε ότι η Τουρκία δεν είναι δημοκρατική χώρα. Για άλλη μια φορά βλέπουμε να υπάρχει θύμος των δημοσιογράφων από το καθεστώς Ερντογάν. Με την Τουρκία μιλάμε για ένα στιμοκρατούμενο κράτος. Ε, σήμερα τίποτα δεν σταματάει τον Ερντογάν. Ε, εκείνος ε, συλλαμβάνει και φυλακίζει. Οπότε, πριν από 10 χρόνια ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Όμως, εγώ ως ε, μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Τουρκία έχω δύο λύσεις να προτείνω. Πρώτα απ' όλα να δοθεί τέρμα στην απελευθέρωση του καθεστώτων των θεωρήσεων και από την άλλη να δοθεί τέρμα σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ε, για ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Πάμπριξ τώρα, λεπτό. Κυρίες και κύριοι, Κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν διάφοροι υποστηριχτέ τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πω ότι όλοι μα ανησυχούμε για τα όσα συμβαίνουν και για αυτά που κάνει η κυβέρνηση στη Τουρκία. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση στη Τουρκία πηγαίνει όλο και περισσότερο προς ε, την κατάσταση αυτή στην οποία πηγαίνει και η Ρωσία. Η Τουρκία ως κράτος, ως κοινωνία, ως κυβέρνηση. Και αν έχουμε αρνητική στάση, όπως προτείνουν ορισμένοι εδώ, απέναντι στην Τουρκία να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις, για παράδειγμα, και οικονομικές κυρώσει. τότε τελικά ένα μεγάλο μέρος πραγματικά ε, Τούρκων οι οποίοι προσανατολίζονται στην ελευθερία και που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες με εμά, τους εγκαταλείπουμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να επηρεάσουμε την τουρκική κυβέρνηση. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα στοχεύσουμε καλύτερα την βοήθειά μας, τη βοήθεια που δίνουμε σε χώρα προς ένταξη. Πήγε η κυρία Μογκερίνη στη Γάζα, θα έπρεπε να δει έτσι και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι Παγώνοντας τα κεφάλαια 23 και 24, στρέφουμε την Τουρκία προς μια πλευρά όπου δεν θα μπορούμε πια να την επηρεάσουμε, ενώ τόσο πολύ χρειάζεται αυτό. Ευχαριστώ κύριο Μποστινάρου τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να επαναλάβουμε κάτι προφανές, ότι η ελευθερία τύπου είναι βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Οι συλλήψεις λοιπόν της Κυριακής είναι απαράδεκτες. Δεν είναι δυνατόν να τις δεχτούμε γιατί αμφισβητεί την ίδια την έννοια της ελευθερίας στην Τουρκία. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία που είναι προς ένταξη χώρα πρέπει να είναι ανοιχτές και ειλικρινείς. Εμείς οι σοσιαλιστές και θέλουμε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένταξη της Τουρκίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και για τα εμπόδια. Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε αντιμέτωποι με την ε, στέρηση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία. Σίγουρα ανησυχούμε για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία και τη στάση του Πρωθυπουργού Ερντογάν. Πρέπει να δείξουμε, για να καταδείξουμε στην Τουρκία τις ευθύνες της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σούλτσε για ένα λεπτό τώρα. Ενάμιση λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, τα γεγονότα στην Τουρκία ε, είναι πολύ ανησυχητικά. Το καθεστώς του Προέδρου Ερντογάν κάνει πραξικοπήματα κατά του τύπου και συλλαμβάνει τους ανεπιθύμητους ε, δημοσιογράφους. Εγώ ως ε, Ανατολικογερμανός ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει έλλειψη ελευθερία του τύπου. Η στάση τη τουρκική κυβέρνηση είναι απόλυτα απαράδεκτη κατά των θεμελιωδών αρχών τη Ένωση. Είναι δυνατόν μια τέτοια χώρα να γίνει ποτέ μέλο τη Ένωση που δεν σέβεται το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ νομίζω όχι. Η δημοκρατία δεν σημαίνει, ότι όλοι πρέπει να πιστεύουμε τα ίδια και μια κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Δημοκρατία σημαίνει το κράτος και η κοινωνία να σέβεται τον πλουραλισμό και την ελευθερία έκφρασης με την φυλάκιση των ε, δημοσιογράφων έδειξε για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο η κυβέρνηση Ερντοάν. Η κυβέρνηση η οποία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη και από κάθε δημοκρατική αρχή. Ξεκίνησε με την βίαιη καταστολή των διαδηλωτών στον Κεζί και συνεχίζεται με αυτές τις κρατήσεις των αντιπάλων του Ερντοάν. Ο Ερντοάν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα δεν θα τον εμποδίσουν σε τίποτα. Η κυρία Μογερίνη και η Κομισιόν πρέπει να αποστείλουν ισχυρό μήνυμα. Η διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η τελευταία ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε, αλλά μπορεί και να χρειαστεί να γίνει. Η τελευταία καταφυγή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Έρτουγκ. Να δούμε λίγο σύντομα την ιστορία. Το Σεπτέμβριο 2005 ήταν ε, το καλύτερο σημείο των σχέσεων μας με την Τουρκία όταν ε, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα πριν από ένα χρόνο είχαμε την ε, μεγαλύτερη περίπτωση διαφθοράς στην Τουρκία όπου χρειάστηκε να παρατηθούν τέσσερις υπουργοί και την περασμένη Κυριακή συνελήφθησαν πολλοί δημοσιογράφοι χωρίς καθόλου ενδείξεις μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν υποψίες. Γι' αυτό Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Τουρκία ήταν ισχυρή μόνο όταν ήταν στραμμένη προς την Ένωση. Για παράδειγμα, από το 5 ως το 11 είχε αύξηση περίπου 6% το χρόνο, ενώ πέρυσι ήταν 3 ε, και κάτι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη γενική οικονομική κρίση. Γι' αυτό κάνω έκκληση προς το καθεστώς να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις και να βελτιώσετε την νομοθεσία σας να προσαρμοστεί προς την νομοθεσία της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέναρς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Τουρκία είναι μια χώρα στην οποία παρατηρούμε διώξεις δημοσιογράφων, άρα δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία Ξέρουμε τι ιστορία έχει στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τηρεί τα κριτήρια. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να σημειώσει. Εννοείται ότι τον Ιανουάριο πρέπει να καταδικάσουμε τις πράξεις αυτές. Δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να αφήσουμε μόνη της τη χώρα αυτή. Ζήτησε η ίδια η Ολλανδική κυβέρνηση σήμερα από το Συμβούλιο να παγώσει τις διαπραγματεύσεις. Άκουσα και τους συναδέρφους τι είπανε ότι πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία της Τουρκίας. Αυτό είναι αλήθεια. Και να τη στηρίξουμε περισσότερο. Οπότε εγώ ρωτάω το Συμβούλιο τι δυνατότητες υπάρχουν να χρησιμοποιήσουμε την πάυση των διαπραγματεύσεων ως πίεση, αλλά από την άλλη μεριά να βοηθήσουμε την κοινωνία της Τουρκίας και τους ανθρώπους εκείνους στην Τουρκία που πιστεύουν στις ευρωπαϊκές αξίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να καταδικάσω την πρόσφατη επιχείρηση φήμωσης του τύπου και ενίσχυσης ελέγχου του διαδικτύου από την τουρκική κυβέρνηση. Οι πρακτικές αυτές πλήττουν τι θεμελιώδει αρχέ ελευθερία του λόγου μα πάνω απ' όλα πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία. έχοντα σταθερά υποστηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική τη τουρκία εκφράζω την ανησυχία μου για αυτή την εξέλιξη η οποία αποτελεί δείγμα οπισθοδρόμηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. αγαπητοί συνάδελφοι πέρυσι είχαμε τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο κέντρο τη κωνσταντινούπολη. πιο πρόσφατα συναντήσαμε την αμφίσιμη στάση τη τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά τον αγώνα του διεθνή συνασπισμού ενάντια στους τζιχαντιστές του Ίσες. μόλις τον προηγούμενο μήνα καταδικάσαμε την παραβίαση της, τη κυριαρχίας της κύπρου ενός κράτους μέλους μας από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και ξανά σήμερα σε ακόμα μία ολομέλεια συζητάμε για ένα νέο πλήγμα κατά της ελευθερίας του τύπου στην τουρκία. δυστυχώς όλα αυτά συνιστούν ενδείξεις ότι ο ερντογάν οδηγεί την Τουρκία μακριά από τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Θεοχάρου για λεπτό. Στις ψευδεσίσεις μερικών η Τουρκία δεν είναι δημοκρατική χώρα. Παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα εκατομμυρίων πολιτών και η ελευθερία του τύπου βιάζεται καθημερινά επιπλέον η τουρκία κατέχει στρατιωτικά τμήμα της κυπριακής δημοκρατίας. οι τελευταίες συλλήψεις τούρκων δημοσιογράφων από το καθεστώς Ερτογάν, που συνεχίζουν ανάλογες πρακτικές του παρελθόντος δείχνει ότι ο Ερτογάν σοβαρομιλούσε όταν έλεγε, ότι θα έλεγε προεκλογικά ότι θα λιώσει όλου όσοι εναντιώνονταν σε αυτόν. Τη προάλλε μα είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να ανακατεύεται με του οίκου του την τουρκία αυτή κανείς δεν τη θέλει στην ευρωπαϊκή ένωση. γι' αυτό πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές συνομιλίες και η προενταξιακή βοήθεια προς την τουρκία μέχρι να αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται την πολιτική ηθική της ευρώπης. οι οικονομικές συναλλαγές με την τουρκία είναι τεράστιες αλλά οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε και τις αρχές και τις αξίες μας που βιάζονται συστηματικά από αυτή τη χώρα. Επιπλέον, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υπερασπιστεί στην Κύπρο τις αρχέ και τις αξίες τη όπω πράττει στην Ουκρανία και όπως κάποιοι είπαν μέσα στην Τουρκία, δεν θα γλιτώσει από την παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λόπες. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και των ατομικών ε, δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ στην Τουρκία. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν αυτό με του δημοσιογράφου την προηγούμενη εβδομάδα. Που αποτελεί μία παραπάνω περίπτωση σε τόσε άλλες που έχουν λάβει χώρα στην Τουρκία, όπου η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο πολύ συχνό που δεν υπάρχει ανεξαρτησία, που υπάρχουν επιθέσεις στον τύπο και βλέπουμε και τους πολιτικούς ηγέτες να πλήττουν και τι πολιτικέ ελευθερίε και τι ελευθερίε του συνεταιρίζεσθε. Εμεί λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να καταδικάσουμε τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία. Πρέπει να έχουμε βέβαια μια στάση θετική, όχι με την κυβέρνηση, αλλά για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το μέλλον της Τουρκίας. Αυτή είναι δικιά μας υποχρέωση. Όχι απέναντι στην κυβέρνηση υποχρέωση, αλλά απέναντι στο λαό της Τουρκίας. Ο κύριος Ρούα τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε τις πρόσφατες ε, συλλήψεις στην Τουρκία και την καταπίεση της ελευθεροτυπίας στη χώρα αυτή που είναι υποψήφια για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κράτος δικαίου και ο δικαστικός κλάδος ε, αλλά και η ελευθεροτυπία είναι τρεις πυλώνες ε, καθοριστικοί για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες που βεβαιώνουν το δίκαιο, τις ελευθερίες και την προστασία των πολιτών μας. Η Τουρκία θα έπρεπε να συμπορφώνεται με αυτέ τις αρχέ αφού είναι υποψήφια προς την προσχώρηση. Για αυτούς του λόγου, ε, κύριε εκπρόσωπο τη Ιταλική Προεδρία, ελπίζουμε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη αυτών των συλλήψεων, γιατί πρέπει να λάβουμε γνώση των συγκεκριμένων κατηγοριών κατά του καθενό από αυτού του πολίτε. Απαιτούμε ένα από τα κράτη που είναι υποψήφια για να γίνει μέλο τη Ένωση να διεξάγει ε, ανακρίσει και έρευνε δικαστικέ ε, ανεξάρτητε με τρόπο διαφανή και πέραν κάθε αμφιβολία. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν ότι ε, αυτά, οι δηλώσει που έγιναν απαράδεκτε για να αποτελέσει μέρο τη ομάδα μα. Ευχαριστούμε, κύριο Χρυστοφόρο, για ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό η τουρκία όλα αυτά τα χρόνια μας απέδειξε ότι ένα πράγμα ξέρει να κάνει σωστά και το κάνει με συνέπεια ότι ξέρει να περιφρονεί διαχρονικά όλα τα ψηφίσματα που εκδίδονται να παραβιάζει συστηματικά και διαχρονικά ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο μέσα στην τουρκία αλλά και έξω από την τουρκία να προκαλεί προβλήματα να είναι ο ταραξίας της περιοχής να έχει επεκτατικές και επιθετικές διαθέσεις προς όλους και όλα αυτά τα κάνει η τουρκία και το απέδειξε και στην πράξη ότι τα κάνει γιατί επεδείχθη ανοχή από όλου. η τουρκία δεν καταλαβαίνει από ψηφίσματα και από συζητήσει και αν μέσα από αυτή τη συζήτηση δεν βγουν κυρώσει και μέτρα που οφείλουμε ω ευρωπαϊκή ένωση να το πράξουμε πρωτίστω για την αξιοπρέπειά μα για την αξιοπιστία μα και για τον αυτοσεβασμό μα θα ξέρετε ότι θα είναι ακόμα μια συζήτηση στι τόσε πολλέ που κάναμε οι οποίε δεν θα έχουν καμία απόδοση. η τουρκία είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στην πράξη να αποδείξει ότι έχει φιλοευρωπαϊκή πορεία εδώ και χρόνια που όχι μόνο δεν το έπραξε αλλά παίρνει μόνο τα λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να κοροϊδεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριο Ερτογάν να μα προκαλεί και να μα λέει ότι να κάνουμε τη δουλειά μα. Ναι, ο μόνο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μα ένα είναι. Σήμερα να αποφασίσουμε και να καλέσουμε την Ευρώπη να πάρει μέτρα και κυρώσεις οικονομικά. Μόνο αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Διαφορετικά κάθε δύο μήνες θα είμαστε εδώ να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Έληξε ο χρόνο σα Αρχίζουμε την διαδικασία Catch the Eye. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω σε κάποια πράγματα που άκουσα από τους Έλληνες συναδέρφους. Ορισμένα είναι ορθά. Αλλά κάποιοι από τους μη γεγραμμένους προσπάθησαν να πιέσουν και να βάλουν τα δικά τους θέματα στην συζήτηση, κάτι το οποίο πιστεύω ότι τραβάει πάρα πολύ την σοβαρή αυτή συζήτηση. Εγώ είμαι φίλος της Τουρκίας, αλλά οι καταχρήσει στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει μόνο τις χώρες εκείνες που έχουν τις ίδιες αξίες με εμά. Και η Τουρκία ως υποψήφια χώρα αξίζει ξεκάθαρα λόγια από το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Κύριε Μαρίτης, παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οι επιθέσεις που οδήγησαν στην ε, σύλληψη 24 δημοσιογράφων και δύο ε, υπαλλήλων της αστυνομία, καθώς και ηθινών των, των τηλεοπτικών καναλιών δεν μπορούν να περνά παρατήρητες. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσουμε από τις τουρκικές αρχές με απόλυτη σαφήνεια να βεβαιωθούν ότι δεν παραβιάζουν τα βασικά ανθρωπινά δικαιώματα και τα ίδια τα δημοκρατικά θεμέλια της Τουρκίας. Η ανεξαρτησία των ε, ερευνών και του δικαστικού συστήματο είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε υγιού δημοκρατία και θα πρέπει να συμβαίνει αυτό και στην Τουρκία. Οι συλλέψει αυτή ε, καταδικάστηκαν από τον κυρία Μογκερίνη και τον κύριο Πιτέλα αντιφάσκουν με την ελευθερωτική και τι αρχέ τη δημοκρατία και δεν έχουν σχέση με τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου φιλοδοξεί να γίνει μέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια δημοκρατική και σύγχρονη χώρα που θέλει να προτίθεται να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το να χωρί μαζικέ συλλήψει είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε, συνάδελφο. Ο κύριο Μαριά. Πρόεδρε, η Τουρκία συνεχίζει τη γνωστή τη τακτική, παραβιάζει βάναυσα τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και των μειονοτήτων. Για άλλη μια φορά εξαπέλυσε πογκρόμ διώξεων κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. επιβεβαιώνεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η χώρα αυτή δεν σέβεται τις βασικές δημοκρατικές αρχές της σύγχρονης ευρώπης όταν όμως ένα καθεστώς δεν είναι δημοκρατικό τότε αυτό εκφράζεται και στην εξωτερική του πολιτική. έτσι η τουρκία διατηρεί παράνομα σε ισχύ το casus belli κατά της ελλάδος στο βαθμό που η πατρίδα μου εφαρμόσει άκουσον άκουσον το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το τελευταίο διάστημα εντελώς παράνομα η Τουρκία πραγματοποιεί σεισμογραφικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΣ της Τουρκία η τουρκία πρέπει να λάβει το μήνυμα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και να κληθεί να αποσύρει άμεσα τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την κύπρο και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. ευχαριστώ. Euh, Υπάρχει γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε. Ωραία. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Απλώς να ρωτήσω τον εξαιρετό συνάδελφο. Δεν θα ήταν καλύτερα αν εμείς η Ευρώπη είχαμε μια πιο σαφή στάση απέναντι στην Τουρκία. Θυμάμαι πόσο καιρό χρειάστηκε η Ελλάδα για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει λάθος εάν δεν ανοίξει κανένα κεφάλαιο και δεν βελτιώσει, δεν επιτρέψει πρόοδο στη σχέση της με την Τουρκία. Η ερώτηση είναι, δεν βλέπετε ότι η ενεργηγός μας συμμετοχή είναι καλύτερη από το να περιμένουμε παθητικά τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Η απάντησή σας σε 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ε, η Τουρκία έχει δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα επί δεκαετίες ότι δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο ούτε τα δημοκρατικά δικαιώματα. Έχει έρθει η στιγμή να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους τέλος δεν μπορεί να ανεχόμαστε να υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα κατοχής στην κύπρο. αυτό είναι ξεκάθαρο. καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης. Συνεχίζουμε το Καστιάι με τον κύριο Παπαδάκη για ένα λεπτό. Κύριε γιατί κάνουμε ότι είμαστε έκπληκτοι με τη στάση της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία κατέχει τη μισή Κύπρο, μια Τουρκία η οποία διώκει τους Κούρδους, μια Τουρκία η οποία αφαιρεί τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα των ίδιων της των πολιτών. Το μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για να ενταχθεί στην Ευρώπη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις αρχές και τις αξίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσης και όχι να έχει την απέτηση να υποκύψει η ευρώπη στις δικές της αρχές. και όταν λέμε για τουρκία μιλούμε για το καθεστώς ερντογάν το οποίο αναδεικνύει τον νεοοθωμανικό του πρόσωπο σε κάθε περίπτωση. θέλουμε την τουρκία στην ευρωπαϊκή ένωση σεβόμενοι όμως τη δημοκρατία τις αρχές και τις αξίες της ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και με συγχωρείτε για την προφορά του όνοματός σας, ο κ. Τζαμάσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Όσοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία δεν εκπλήσονται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφορα, δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται, Αυτά όλα είναι πρακτικές ενέργειες του καθεστώτος Ερντογάν και τη τουρκική κυβέρνηση. Να σα θυμίσω ότι μιλάμε για ένα ακόμα νέο Οθωμανικό θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα παλιά τη σύνορα. Στηρίζει τη Χαμάς, την Παλαιστίνη. Στηρίζει το Ισλαμικό κράτος στην Συρία και στο Ιράκ. Τι να περιμένουμε από τον Ερντογάν και τον ε, Νταβούντογλου. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης. Ε, ναι, εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την πιθανότητα κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά μιλώ και ε, προς μεγάλη μου δυσαρέσκεια για την Τουρκία. 27 ε, άτομα συλλήφθησαν σε 13 πόλεις σε μια ε, επιχείρηση που ε, οδήγησε στους ε, σε σύλληψη πολλών αντιφρονούντων και επικριτών του καθεστώτος Ερντογάν. Ε, ο κύριος ε, πολλοί, μάλλον ηθήνοντες καναλιών συνελήφθησαν γιατί τόλμησαν να εκφράσουν απόψεις κατά του Ερντογάν. Όμως εναλλακτικέ φωνές κατά της κυβέρνησης θυμώνονται στην Τουρκία. Η ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης στη χώρα αυτή εξαλείφεται και περνάει στον Ισλαμιστικό χώρο η Η επιλογή μα ε, στην Τουρκία φαίνεται να μην υπάρχει πια. Δεν υπάρχει επιλογή προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε καν για το κράτο δικαίου. Πόσο καιρό θα περιμένουμε, συνάδελφοι, συνάδελφοι πριν ε, του κάνουμε να υποστούν τι συνέπειε και να δώσουμε τι απαραίτητε απαντήσει. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μαυρίδη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ένα λεπτό θα κάνω μια σύντομη ανάλυση. Σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία που λέει ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφή επιτέλους μήνυμα στην Τουρκία, απαιτώντας συγκεκριμένα πράγματα, και η άλλη προσέγγιση που λέει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μια επαφή με την Τουρκία, ανοίγοντας της κάποια κεφάλαια, δίνοντας της χώρο. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, και απευθύνομαι και προς την Επιτροπή, δεν έχει τόση σημασία το τι νομίζουμε εμείς εδώ, αλλά πώς αυτό ερμηνεύεται από τον ίδιο τον Ερτογάν στην τουρκία. οι κινήσεις οι καλές προθέσεις το άπλωμα του χεριού από εμάς ερμηνεύεται ως ανταμοιβή από τον Ερτογάν ενώπιον της κοινής του γνώμης. δηλαδή διοχετεύουμε με δύναμη ένα αυθαίρετο καθεστώς. αν είναι αυτό που θέλουμε να το πούμε. αν όχι να πάρουμε την πρώτη επιλογή με αυστηρά μέτρα. σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Καπούτο για να ολοκληρώσουμε το ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Αυτή η θύελα συλλήψεων δημοσιογράφων είναι ένα χαρακτηριστικό παραδείγμα της ε, κυβέρνηση τη Άγκυρας και ε, ουσιαστικά ενισχύει τους αντιφρονούντες. Είναι μια παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών και της δημοκρατίας. Αντίκυνται στα πρότυπα και τις αξίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, την οποία φιλοδοξεί να γίνει μέλος η Τουρκία. Είναι απαράδεκτο μια δημοκρατική χώρα, σύγχρονη χώρα, που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, να προχωρά σε μαζικές συλλήψεις δημοσιογράφων ε, και ηθινόντων των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Πάνω από 70 δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή και πολλοί από αυτού είναι Κούρδοι γιατί κατούνται για λόγου τρομοκρατία, για τρομοκρατικέ ενέργειε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται σεβαστό το απαραβίαστο δικαίωμα στην ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα και εκδίκαση των υποθέσεών του. Είναι θλιβερά όσα συνέβησαν στην Τουρκία και είναι όλα οδεύουν στην σφαλμένη κατεύθυνση μακριά από την Ευρώπη. Αυτή η πορεία μπορεί να φέρει αρνητικέ και σοβαρέ συνέπειε στην Τουρκία για την οικονομική και πολιτική τη συνεργασία με την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε με πυγμή να αντιδράσει και να καταδικάσει. Ε, Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε το Κατστιάι και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντελαβέντοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους βουλευτές που πήραν το λόγο και συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για το εύστοχο των παρεμβάσεων και των επιχειρημάτων που ανέπτυξαν, για τις ανησυχίες που ακούστηκαν. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι ανησυχίες που όλοι συμμεριζόμαστε. Ήταν σκόπιμο να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να σημειώσουμε τις σοβαρότατες ανησυχίες ε, για τα πρόσφατα γεγονότα και να σχεδιάσουμε τη δική μας τοποθέτηση χωρίς καμία αμφισημία και με απόλυτη σαφήνεια και συνοχή να απευθυνθούμε στους Τούρκους συνομιλητές μας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης με τη μέγιστη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να προάγει την ελευθερία της έκφρασης, της ε, ένωσης και της ε, έκφρασης ε, στο διαδίκτυο και εκτός, διότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς αυτά τα δικαιώματα. Η Τουρκία είναι ένας προνομίωχος εταίρος μας, με τον οποίο διαπραγματευόμαστε την αντεχόμενη προσχώρησή του. Θα πρέπει λοιπόν να επικοινωνούμε μαζί τους με απόλυτη εντυμότητα και ειλικρινή. Όπως είπε ο πρόεδρος Σούλτς, η συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες θα πρέπει να είναι ειλικρινής και ανοιχτή. Θέλω Απλώς να θυμίσω μεταξύ των όσων ε, στη συζήτηση αυτό που υπόθηκε για τις χρηματοδοτήσεις. Είναι απλώς μια παρατήρηση στην οποία αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τον τουρκικό προπολογισμό αλλά με κυβερνητικέ οργανώσει και φορεί που πράγουν το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω κατά κύριο λόγο δύο εργαλείων, το μέσο πρωταξιακή βοήθεια και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η μορφή παρέμβαση και υπογραμμίζω μεταξύ άλλων ότι η ανακεφαλή ε, κατανομή απονομή κονδυλίων στην Τουρκία είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των υποψηφίων χωρών. Ως προς την διεύρυνση, ε, σωστό είναι ότι για να υπάρξει εμβάθυνση στις σχέσεις μας και εδραίωση των μεταρρυθμίσεων πρέπει να συνεχιστεί. Ε, η υπεραιτέρω δέσμευση στο κεφάλαιο 3 θα ήταν μια σημαντική ενθάρρυνση. Έχουμε ήδη κάνει πολλά για να ε, εντείνουμε την δέσμευση της Τουρκίας υποψηφίου χώρας και εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτήν την πορεία να εξακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έληξε η συζήτηση.